Παρακαλώ καθίστε, διότι θα ξεκινήσουμε άμεσα τις ψηφοφορίες. start watching with if I can't implement. Do I will have to? I mean, we can. Yeah, no, I just give it the floor to her. Okay, now we start the voting. Πολύ ωραία, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας και να τις έχετε βάλει στα μηχανήματα, ώστε να δώσω το λόγο στην κυρία Κάμερεβερτ η οποία θα μας βοηθήσει στο πρώτο κομμάτι των ψηφοφοριών επειδή πρόκειται για ένα σχέδιο έκθεσης των δύο επιτροπών έμπλε και ΚΑΛΤ. Έχετε το λόγο κυρία Κάμερεβερτ. Υπάρχει πρόβλημα? Ja, vielen herzlichen Dank. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συνεδριάσουμε από κοινού και να ψηφίσουμε επί αυτών των δύο εκθέσεων. Το χωρίσαμε λίγο. Εγώ θα συντονίσω την ψηφοφορία για το Europass και η συνάδελφος Ουλσκοκ θα ε, συντονίσει την ψηφοφορία για το θεματολόγιο δεξιοτήτων. Για τη δική μου ψηφοφορία ο κατάλογος ψηφοφορία καταρτίστηκε βάσει της πρακτικής που ακολουθούμε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Διαφορετικά έγιναν τα πράγματα στην επόμενη ψηφοφορία βάσει των όσων ε, συνηθίζεται να γίνονται στην Επιτροπή Απασχόληση. Επειδή λοιπόν οι δύο κατάλογοι ψηφοφορία είναι κάπω διαφορετικοί, μην ε, αναρωτηθείτε. Υπάρχουν κάπω λίγο διαφορετικέ παραδόσει ε, ανάμεσα στι δύο επιτροπέ. Θα τα καταφέρουμε όμω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις εισηγητές των δύο εκθέσεων, όλους τους ε, σκιώδεις, τις δύο γραμματείες των δύο επιτροπών για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν για το Europass, ε, υποβλήθηκαν 318 τροπολογίες, 36 συμβιβασμοί εξευρέθησαν και θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε να περάσουμε κατευθείαν στη ψηφοφορία ή αν θα ήθελαν οι εισηγητές να λάβουν σύντομα το λόγο. Φαίνεται πως όχι, επομένως μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με την, με την συμβαστική πρόταση 19, υπέρ. 18, 18, με συγχωρείτε. Προτρέχω, ξέρετε. 18, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ Geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 27 κατά, με συγχωρείτε, ήταν αρκετά σαφής η διαφορά. 164-165 που ταυτίζονται, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 166-167 ταυτίζονται, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 173. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, 484 και 485 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 185. Υπέρ. 185. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Καλύτερα όμως να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 47 κατά απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να επαληθεύσουμε. Παρακαλώ. Όχι, όχι. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ επί της τροπολογίας 188. Geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 34 υπέρ, 37 κατά. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189. Ναι, αν θέλετε βεβαίως να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, κανένα πρόβλημα. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε τις προφορίες. Α, με συγχωρείτε. Πραγματικά είχα άλλη εικόνα από εδώ πάνω. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Περνάμε στην 190. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, καλύτερα να υπαλληθεύσουμε. Ψηφίστε για την τροπολογία 19, έναρξη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 33 υπέρ, 41 κατά. Πρέπει να συνηθίσω το ότι είμαστε μαζί και οι δύο επιτροπέ. Ίσως γι' αυτό κάνω λάθος. Στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού τα πράγματα έχω καλύτερη εποπτεία του τι συμβαίνει. Με συγχωρείτε. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 197 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 198, 199 και 200 που ταυτίζονται υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, ξανά υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε τη 39 υπέρ, 35 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 204 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Επαλήθευση λοιπόν, ψηφίστε, ένας ψηφοφορίας. Geschlossen. Πέραση της ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 34 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 23 και την 216 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν ήταν πολύ σαφές. Ψηφίστε παρακαλώ επί της 224. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 44 υπέρ 27 κατά. 24, 227, 225, όλες μαζί επειδή ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226, απεσύρθη. Πάμε στη συμβαστική 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 28. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. 246, 245, 246 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 36 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται λοιπόν. 249 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 252 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 253, 254, 255 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 256 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 257 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 258 υπέρ, κατά, αποχές, Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Για την τροπολογία 258. Πέρας. 41 υπέρ, 32 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Περκατά κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28, 265, 266. 267, 268. Όλες αυτές ταυτίζονται υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 273 υπέρ Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. 2,75. Περ, κατά, ποιες. Καλύτερα να το επαληθεύσουμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 34 κατά, εγκρίνεται. 276 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286, 287 288, 289, 285 ταυτίζονται υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 299, 300, 301, 302. Όχι. Ξαναπάμε πίσω. 293. Νόμιζα ότι το κάναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα 299, 300, 301, 302. Ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 309 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 32 και την 317, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ κα... Συγγνώμη, συγγνώμη. 326. Περνάμε στην 326. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 και 327 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 334 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 354. Στην μεθεπόμενη σελίδα. 354. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 355. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 356. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 στην επόμενη σελίδα. 58 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 4, συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 63, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Περνάμε στην τροπολογία 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 930, mhm. 131. 9, 130, 131, 132 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 133 υπέρ, κατά, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, έπρεπε να είχαμε περάσει στην 135, έχετε δίκιο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. 144. Υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. 146. Υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 69 υπέρ, 4 αποχές, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές και έχουμε και μια δεύτερη ψηφοφορία να κάνουμε για την εντολή διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο και αυτό θα το κάνουμε ονομαστικά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίστε Χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση. Ψηφίστε παρακαλώ. Abstimmung ist geschlossen. 64 υπέρ, 6 κατά, 2 εποχές. Υπάρχει λοιπόν απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη απόσταση, συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία σε διαπραγματεύσει ο λόγος στη συνάδελφο Μαρίτα Ούλσκοκ για την επόμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε με τη δεύτερη λίστα ψηφοφοριών, ξεκινώντας με την τροπολογία 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, η 113 καταπίπτει, α όχι δεν καταπίπτει, όποιος είναι υπέρ της 113 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 114 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 55 ψήφους τροπολογία 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Να ελέγξουμε την 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 46. Συμβιβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική ε. Στη σελίδα 3. Υπέρ κατά αποχές συμβιβαστική ε σελίδα 3 επαναλαμβάνω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και μετά πάμε στην συμβιβαστική QA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 127 στη σελίδα 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 131 έως η ΙΝΚΟ 7 καταπίπτει. Και πάμε στη συμβιβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία... ...145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται μάλλον... ...να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 145. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με κατά, τρεις ψήφους παραπάνω. Τροπολογία 146 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 148 Ψηφίζουμε την 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 148 για να είμαστε βέβαιοι. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 6 ψήφους παραπάνω. Τροπολογία 140, 150, συγγνώμη. Συγγνώμη, 149. 150. υπέρ κατά αποχές ε, δεν βλέπω δεν φαίνεται τα χέρια σας ξαναρχίζουμε 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 154 ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 43 ψήφους. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 159. Ζητά συγγνώμη πρόεδρος. 158 θέλετε να ελέγξουμε, λέτε. Ωραία, να ελέγξουμε το 158. Τροπολογία 158. Ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας για την τροπολογία 158 εγκρίνεται με 42 ψήφους 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά δύσκολο δεν φαίνονται τα χέρια σας ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 162 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 162 ηλεκτρονικά, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 67 ψήφους. Μόνο πέντε όμως σηκώστε τα χέρια σας. Άντε οκτώ. Τροπολογία 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1.65 καταπίπτει. Συμβιβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 171. Στην επόμενη σελίδα. Είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 171. Άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, Απορρίπτεται. Τροπολογία 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Συμβιβαστική συγγνώμη W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβαστική συγγνώμη H. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 178. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας για την 178. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Τροπολογία, για να δούμε τώρα. «183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική κάπα, στην ίδια σελίδα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 188. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 189, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 90, όχι, συγγνώμη, 91, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 193 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει και πάμε στην 194. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 195 ε, προφορική τροπολογία όχι ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας ποιος είναι κατά αποχές εγκρίνεται 196 ποιος είναι υπέρ ποιος είναι κατά αποχές εγκρίνεται. 198 επίσης προφορική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο Λάθος. Συμβαστική J είναι η επόμενη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική L. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 209. Υπέρ, ε, κατά, να ελέγξουμε την 209. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 62 ψήφους. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 219 ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κα, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα Το θέτουμε ναι. δεύτερο τμήμα της 19 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 2.20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.21 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Αψηφίζουμε για αυτήν. 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2.33 πρώτο τμήμα 2.23 συγγνώμη ε, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε την 2.23 το άρχεται ψηφοφορία το δεύτερο τμήμα της 2.23 δεύτερο τμήμα της 2.23 και πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με, κατά τέσσερις ψήφους 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 θα ψηφίστε υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 230 Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Τελευταίο τμήμα της 2.30. Δεύτερο τμήμα, τελευταίο τμήμα της 2.30. 2.32, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, δεν βλέπω, πρέπει να ψηφίσουμε. Τελευταίο τμήμα της 232, άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους. 226. vote on the last, but I mean, you voted on that, we adapt. Yeah. Okay. Okay. It's to be voted those in favor, those against. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 2.27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.34 κατά πρέπει να ψηφιστεί υπέρ της 2.34 κατά της 2.34 απορρίπτεται να ελέγξουμε τη 2.34 με ηλεκτρονική ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 10 ψήφους παραπάνω, 2.35 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.28 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 2.30 κατά καταπίπτει Πάμε στην 2.46 στη σελίδα 22. 2.46 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 2.46. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 247 ηλεκτρονικά. Άρχεται, πέρας, εγκρίνεται με 50 ψήφους. 2.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.48 Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.51 Καταπίπτει, πάμε στην 2.52 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.55 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε τη 255 Έρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται κατά μία ψήφο 253 υπέρ είναι συμβατή όχι ε, λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 καταπίπτει 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι να την ελέγξουμε 264 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 46 ψήφους. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 269. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 269 άρχεται ψηφοφορία πέρα ψηφοφορία, εγκρίνεται με 52 ψήφους τροπολογία 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ανθρωπολογία 2.77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.79 συγγνώμη 2.80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 281 και 282 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την 283 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται θα έλεγα. 285 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 285 άρχη η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 64 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 288 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 289 we να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Yeah. That was the result. Uh, and now we have mm-hmm. 290. 290, yes. Amendment 290, those in favor. 290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική νη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε μετά στην ΙΜΚΟ 11. Δεύτερο τμήμα στη σελίδα 27 υπέρ κατά αποχές να το ξαναδούμε ΙΜΚΟ 11 υπέρ πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται Προπολογία 300, 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 300. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 45 υπέρ. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πι Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν τώρα στην 315 στη δική μου σελίδα σε 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά εγκρίνεται 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 332 Στη σελίδα 32 υπέρ 332 κατά αποχές εγκρίνεται για την 332 ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται πέρας εγκρίνεται 35 λοιπόν και 30 5 υπέρ 334 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Την 3.35 θα την κοιτάξουμε, ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3.43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.47 υπέρ, κατά, αποχές, Πρέπει να το δούμε ηλεκτρονικά, γιατί 347 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 38 με 32. 342 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 350 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 358 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 363 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 375 υπέρ στη σελίδα 37 κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη, οπότε θα το δούμε ηλεκτρονικά. Στην 375 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 40 με 23. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η συμβαστική R υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. «389». Σελίδα 39 για μένα. Στην 389 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3,90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3,91 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 3,92 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 3,93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3,94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 395 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. Υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα δεκατρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα δεκατέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα δεκαπέντε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 416 υπέρ καταπίπτει οπότε πάμε στη 17 υπέρ 417 κατά αποχές απορρίπτεται Τέσσερα εικοσιένα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 418 ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής απορρίπτεται 419 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4.25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4.26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Για την 4.26 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 33-43. Ήμκο 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική X Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά συμβιβαστική Y Στη σελίδα 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.45 στη σελίδα 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 447 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 449 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 449. Άρχεται, πέρας, απορρίπτεται. 63 με 12. 4,50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 4,51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 4,52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, την 452 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 39-31. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 454 καταπίπτει.

υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 457 υπέρ κατά τη 456 λοιπόν παρακαλώ ηλεκτρονικά άρχεται Συγγνώμη, την 457 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, την 457 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 36-44, λοιπόν ε, περισσότερες ψήφοι κατά και μετά 4-59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4-60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4-64 υπέρ κατά α, αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ ή μάλλον όχι 464 υπέρ διανατάσεως κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 472 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,77 υπέρ. Α, λοιπόν. 476 ηλεκτρονικά. Επανερχόμαστε. 476 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 477 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 474 Καταπίπτει. Τέσσερα εβδομήντα οκτώ υπέρ. Okay, we have to vote on 478. Those in favor? Περ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 479. Καταπίπτει. 480 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 481 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά μπορούμε την 481 να τη δούμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται πέρας Κατα... Ε, ε, απορρίπτεται. 482 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 483 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 484 υπέρ. Κατά εγκρίνουμε τη 484 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. 72 υπέρ. 4,87 είναι η επόμενη. 487 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 488 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 489 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 490 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 491 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 492 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 493 υπέρ κατά αποχές. Για να δούμε την 493 λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 494 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 496 καταπίπτει 497 497 υπέρ κατά αποχές νούμερο εγκρίνεται 498 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 499 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται 500 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά την 500 παρακαλώ Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 501 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 502 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 503 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 504 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 505 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 506 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 507 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θα ψηφίσουμε την 508, 508 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 509 καταπίπτει, η επόμενη που ψηφίζουμε είναι η 511, 511 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 512 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 5.13 υπέρ, κατά, χέρ, απορρίπτεται, ημκο 1 υπέρ, κατά, Οι τέσσερις της ημκο μαζί, 1, 2, 3 και 5. Θέλετε να τις κάνουμε μία-μία υπέρκατα τις της 1 αποχές να το δούμε so that we know the rest. The vote is closed. Άρχεται πέρας εγκρίνεται ΙΜΚΟ δύο υπέρ αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές. Η μία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νούμερο 2 υπέρ κατά υπέρ εποχές με συγχωρείτε απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20, η 20 καταπίπτει, η 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, οι 6 και η 7 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 9 διαγράφεται, υπέρ λοιπόν της διαγραφής, κατά,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 αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κα... υπέρ πάλι για την 26 υπέρ και τώρα κατά ωραία ευχαριστώ απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ την 27 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται λίγη. Πολύ δύσκολη αυτή. 28. Η κυρία Γιασλοβίτσκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ, Σον Σάιμον. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται.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 αποχές. Για να δούμε το δεύτερο τμήμα της 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να το δούμε ηλεκτρονικά, να δούμε τη 43 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές να το δούμε λοιπόν τη 49 The vote is open and the vote is now closed. Yes, 72 votes. Άρχεται και ναι με 42 εγκρίνεται. Περνάμε στη 50 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 και 54 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές για να δούμε το 57 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας Λοιπόν, απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. You want to check amendment 15? Θέλετε να ψηφίσουμε για την 59. Ψηφίστε. Πέρασε τους προφορές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Να ψηφίσουμε για την 68. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44 υπέρ, 30 κατά. Με συγχωρείτε. 69 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ε, απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. «73 δεν σηκώθηκε σχεδόν ούτε ένα χέρι» στην αίθουσα. Πάμε ξανά. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Γιατί δεν ήταν σαφές. Ψηφίζουμε την τροπολογία 73. Τέλος της ψηφοφορίας. Oh, there was some mistake with the, the machinery. We make it once again. Υπήρξε ένα ασφαλό με το μηχάνημα. Ξανά. Τροπολογία 73. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με διαφορά 7 ψήφων. Σεβαστική Β. Υπέρ. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Εποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Και περνάμε στην 90 υπέρ κατά ποιες ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 91. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Κρίνεται. 51 ψήφους υπέρ. 92 υπέρ. τα Ποιες. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. τα Ποιες. Απορρίπτεται. Καλύτερα να ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά για την τροπολογία 95. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε τις προφορίες. It's rejected by seven votes. Amendment 98, those in favor. Πάμε στα επόμενα 98 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Ποιες απορρίπτεται να ελέγξουμε. Για την 101 ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Τα Αρχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Τα Ποχές Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 62 κατά. 109 καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 96 και 110 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, ποιες εγκρίνονται. 104 μαζί με την 111 που επίσης ταυτίζονται υπέρ, τα, εγκρίνονται εγκρίνονται. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε τώρα επί της έκθεσης στο σύνολό τη. Ονομαστικά, ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε στις οφορίες. 59 υπέρ. Ευχαριστούμε τη Μαρτίνα Τλαβαγιώβα για τον Μόμτσιλ Νέκοβ για το έργο τους, για την έκθεσή τους με θέμα το